που αναφέρθηκε χθε στην χθεσινή συνεδρίαση δεν εκφράστηκαν σχετικέ ενστάσει εντό 24 ώρων και σύμφωνα με τον κανόνα 105 παράγραφο 4 εγκρίνεται η σύσταση. Αυτή θα δημοσιευτεί με τα εγκεκριμένα κείμενα αύριο ε, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου του 2014. Να ενημερώσω επίση το Κοινοβούλιο ότι σύμφωνα με τον κανόνα 231 παράγραφος 4